Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτήν την τραγική ανακοίνωση θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν ήδη μοιραστεί, υπάρχουν παρατηρήσεις από αυτόν. Δεν βλέπω, επομένως θεωρούνται εγκεκριμένοι.